για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Φέρβερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, ε, στην Ευρώπη οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ε, συμβάλλουν σημαντικά στην συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2007 έχουμε, είχαμε την ε, τρίτη οδηγία, τη διαπραγματεύτηκα και εγώ και τότε λοιπόν πραγματικά μας ενδιέφερε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την συνοχή και τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Τότε είχαμε ταχυδρομικές υπηρεσίες που ακολούθησαν μια πολύ καλή κατεύθυνση, είχαμε ανταγωνισμό. Ε, μέσα στα κράτη-μέλη είχαμε νέους ε, παρόχους ε, και εμφανίστηκαν και άλλοι καινούργοι στην αγορά ε, διαδόθηκε λοιπόν η προσφορά, πήγαν όλα μια χαρά. Βεβαίω με την ε, ψηφιοποίηση τη επικοινωνία κατά τον 21ο αιώνα είχαμε και ριζικέ αλλαγέ και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρέπει όμω να έχουμε κατά νου ότι οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε, οι οποίε πριν από 10 χρόνια εμφανίστηκαν ε, πολύ ενεργά στην ευρωπαϊκή αγορά τώρα αυτέ πλέον αποσύρθηκαν σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Εμεί δεν τη θέλαμε αυτή την εξέλιξη. Εμείς θέλαμε περισσότερο ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα τελειώσω με μια, ένα παράθεση από τον Βολτέρο που είπε το ταχυδρομείο παρηγορεί τον άνθρωπο, είναι η παρηγοριά του ανθρώπου γιατί μετατρέπει τους απόντες σε παρόντες. Τέλος της παράθεσης του Βολτέρου. Καλύτερο από αυτό δεν μπορούσα να βρω. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ήδη από ε, τη δεκαετία του 90 είχαμε ε, συμφωνήσει με τον κύριο Μπράνι Σίμψον που ήταν ο πρώτος εισηγητής ε, της ε, πρώτης οδηγίας για τις αρχιδρομικές υπηρεσίες το 1997. Τότε είχαμε μιλήσει για καθολικές υπηρεσίες γιατί τότε μας ενδιέφερε πάρα πολύ όχι μόνο οι άνθρωποι στις αστικές περιοχές να έχουν καλές ταχυδρομικές υπηρεσίες αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές στα βουνά, στα νησιά, στις περιφέρειες, στις ε, απόκεντρες λίγο περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι να είναι προσπελάσιμοι με ταχυδρομικές υπηρεσίες. Μετά από 10 χρόνια διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη και ε, με έκπληξή μου διαπίστωσα ότι έχουμε ένα κράτος μέλος όπου το 25% του πληθυσμού, μεγάλο μάλιστα κράτος μέλος, ε, που έχει πει ότι δεν χρειάζεται να στέλνονται κάθε μέρα γράμματα. Αυτό δεν είναι στο πλαίσιο αυτού που είχαμε είχαμε συμφωνήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι οι πάροχοι καθολικών υπηρεσιών θα πρέπει να ε, λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο και αυτό ισχύει μέσα από την απαλλαγή από το ΦΠΑ. Και θέλω να σας επισημάνω ότι όσοι έχουμε καθολικές υπηρεσίες έχουν ένα εργαλείο το οποίο δεν έχουν οι ανταγωνιστές τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι και προς το δικό μας συμφέρον όσοι έχουν αυτό το προνόμιο προνόμιο της απαλλαγής ε, ΦΠΑ, ε, από ΦΠΑ των ε, ταχυδρομικών υπηρεσιών, των γραμματοσύμων, αυτή να είναι πιο ανταγωνιστική. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για ταχυδρομικές υπηρεσίες, για μεγάλους μικρούς παρόχους, ε, όπως και για διασυνοριακές υπηρεσίες. Επιθυμούμε οι υποπτικές αρχές να μεριμνήσουν έτσι ώστε να υπάρχουν εχέγγυα και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στις εθνικές αρχές έτσι ώστε και οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ θερμά κυρίως ε, τις σκιώδεις εισηγήτριές μου και τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύ επικοδομητική συνεργασία. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα ε, γιατί από τότε, από την ομάδα του 2007 έχω μείνει μόνο εγώ. Αλλά τελικά εντάξει Εντάξει, καλά τα καταφέραμε και χαίρομαι για τη συζήτηση και ελπίζω αύριο να εκπέμψουμε ένα σαφές μήνυμα για ισχυρές καθολικές υπηρεσίες που τα προσφέρονται στους πολίτες μας. Ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση διας πρωτοβουλίας ε, και ιδιαίτερα τον κύριο Φέρμπερ και τους ε, εισηγητές των επιτροπών που γνωμοδότησαν. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίε είναι σημαντικός τομέας της ε, οικονομίας. Το 2014 πάνω από 500 εκατομμύρια δέματα και πακέτα και 64 δισεκατομμύρια επιστολές εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ο κλάδος αυτός ε, αλλάζει. Την ίδια χρονιά ο αριθμός των επιστολών που εστάλησαν είχε μειωθεί κατά 4%. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, μάλιστα, οι μειώσει ήταν ακόμα σημαντικέ, πιο σημαντικέ. Στη Δανία ήταν 14% η μείωση, ενώ στην Ιταλία ήταν πάνω από 9%. Από την άλλη μεριά, ο αριθμό των δεμάτων και των πακέτων αυξάνεται ταχύτατα εξαιτία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η βελτίωση του διασυνοριακού εμπορικού, ε, ηλεκτρονικού εμπορίου είναι στοχο τη ε, ε, ψηφιακού μα προγράμματο ε, θα επανέλθω στα δέματα βέβαια, αλλά να πω δύο λόγια για την οδηγία ε, ταχυδρομικών υπηρεσιών. Όπως ξέρετε, ε, υιοθετήσαμε την ε, έκθεσή μας για την εφαρμογή της οδηγίας στο τέλος του περασμένου χρόνου και το συμπέρασμα ήταν ότι χρειάζεται περισσότερη ανάλυση και ότι κάθε χρόνο θα δημοσιεύουμε στατιστικά. Έχει, μπορώ με χαρά να σας πω ότι τα τελευταία στατιστικά για το 2014 δημοσιεύθηκαν στο site μας των, της Κομισιόν τον Ιούνιο. Επίση, δημιουργούμε μια ομάδα εργασία για τα στατιστικά των χειδρομικών υπηρεσιών. Ε, προσπαθούμε να αυτοματοποιήσουμε τη συλλογή πληροφοριών για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να επιταχύνουμε τη δημοσίευσή του. Η οδηγία ταχυδρομικών υπηρεσιών απαιτεί σε αυτόν προσφέρει καθολικέ καθολικές να ε, παραδίδει πέντε μέρε τη βδομάδα και δέματα και επιστολέ εκτό εξαιρετικών περιπτώσεων. Όμω οι ε, πολίτε μετακινούνται σε πιο ηλεκτρονικέ μορφέ ε, επικοινωνίες, οπότε ε, γίνεται πολύ πιο ακριβή η επίδοση κάθε μέρα. Για παράδειγμα, οι επιστολέ τριών γραμμάτων, η επίδοσή του αυξήθηκε η τιμή τη κατά 7,5% πέρσι. Χρειάζεται λοιπόν ευελιξία για το πώ τα κράτη-μέλη θα εφαρμόζουν την οδηγία ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αυτό θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν στις αλλαγές των συνηθιών των ε, πελατών. Ε, τώρα, λιγότερα κρατή μέλη ε, συμπεριλαμβάνουν τις εφημερίδες στις καθολικές υπηρεσίες ενώ, κάποιες, ενώ λίγες χώρες επιμένουν σε 6 μέρες αντί στις 5 μέρες επίδοση κάθε εβδομάδα οι, οι ταχυδρομικές πίεσεις, καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες θα μπορούν να επιδοτούνται, αλλά θα πρέπει οι επιδοτήσεις να περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο ε, και να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Ε, στην ε, έκθεσή μας αναφέρουμε και, μια, και μεθόδους υπολογισμού των επιδοτήσεων που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλες. Η έκθεσή μας επίσης αναγνωρίζει τον ε, ρόλο των, ε, των εποπτικών ανεξάρτητων ε, ρυθμιστικών αρχών. Το 2010 δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για να, για να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και μάλιστα έκανε πολύ καλή δουλειά αυτή η ομάδα εργασίας. Η ομάδα θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην εφαρμογή της πρότασης ε, για ε, κανονιστικές ρυθμίσεις. Τώρα, επιστρέφω στην επίδοση των δεμάτων. Η πρόταση αυτή οθετήθηκε το Μάιο ως τμήμα του πακέτου μέτρων για την βελτίωση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Στόχος είναι αλλαγές εκεί που οι αγορές και ο ανταγωνισμός δεν έχουν λειτουργήσει. Ε, σύμφωνα με τον δικό χάρτη του 2013, ε, θέλουμε ε, οι καθολικές υπηρεσίες να είναι διαλειτουργικές. Ο κανονισμός προτείνει δράσεις σε τρεις κυρίως άξονες. Πρώτον, ε, οι ε, κανονιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν πληροφορίες για όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που είναι εγκαταστημένες στα κράτη-μέλη εκτός των μικρότερων. Αυτό θα, τους, θα τις διευκολύνει να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αγορές. Δεύτερον, ε, οι τιμές των ε, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να θα γίνουν πιο διαφανείς. Τρίτον, ε, πρόσβαση στις καθολικές, στα δίκτυα των παρόχων καθολικών υπηρεσιών από τρίτα μέρη χωρίς διακρίσεις. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις μικρές επιχειρήσεις ε, ε, να ε, εξασφαλίζουν καλύτερους κανόνες και όρους. Οι πάροχοι καθολικών υπηρεσιών επίσης θα υποφεληθούν από τον αυξανόμενο αριθμό πακέτων και αυτό θα οδηγήσει σε διατήρηση των θέσεων ασίας ιδιαίτερα στις παραμεθόρες και μεθόρες περιοχές. Τέλος, όπως αναφέρεται στην έκθεσή σας, στην η έκθεση της, όπως αναφέρει η έκθεση Επιτροπής Απασχόλησης, η ε, οδηγία ταχυδρομικών ε, υπηρεσιών ε, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη τη, τους εργασιακούς κανόνες στην αδειοδότηση. Μπορούν να απαιτούν δηλαδή κάποιες ελάχιστους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω να ακούσω τα, τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μάρκου Φέμπα για την έκθεσή του. Για μένα υπάρχουν τρία πράγματα που είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ο κύριο Φέμπερ το έχει ήδη αναφέρει. Ε, να διατηρήσουμε τι ε, καθολικέ υπηρεσίε, τη μορφή που έχουν. Δεύτερον, να επεκταθεί ο ρόλο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Και τρίτον, οι επιπτώσει στου εργαζόμενου να μην αγνοούνται. Γίνονται αλλαγέ και αυτέ έχουν επιπτώσει στου εργαζόμενου. Οι κλασικοί πάροχοι είχαν κατορθώσει να εκπαιδεύσουν καλά τους εργαζόμενους. Ε, ε, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφορές στις συνθήκες εργασίας. Ε, έχουμε ε, επισφαλείς συμβάσεις, ε, αυξάνονται αυτές όλο και περισσότερο. Για μας λοιπόν, για την Επιτροπή Απασχόλησης, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι θα εξακολουθούν να απολαύουν καλών συνθήκων εργασίας, ασφάλεια και κανόνες υγιεινής στην εργασία. Και επίσης να είναι ικανοποιητική και η αποζημίωσή τους. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ καλή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στο μέλλον δεν θα πρέπει να μετακυλείται στους ώμους των εργαζομένων. Κύριε Άντερσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την εκθέση αυτή εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρμπερ και όλου του συναδέλφου από όλε τι επιτροπέ που εργάστηκαν σκληρά. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντικέ αλλαγέ στι ταχυδρομικέ υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την ραγδαία αύξηση του αριθμού των δεμάτων. Η αναθεώρηση τη οδηγία ταχυδρομική υπηρεσία ε, είναι ευκαιρία να αξιολογήσουμε τι αλλαγέ και να καθορίσουμε προτεραιότητε για το μέλλον η, η αναθεώρηση της οδηγίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και η αυριανή ψήφος επιβεβαιώνουν ότι η οδηγία δεν απαιτεί την ιδιωτικοποίηση των, της παροχής καθολικών υπηρεσιών. Ε, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα ε, μιας ε, προσιτής και συνεχούς ε, παροχής υπηρεσιών, καθολικών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ε, επίσης τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να προστατευθούν ε, καθορίζοντας ελάχιστες ε, προδιαγραφές ε, ενώ δίδεται και επαρκής ευελιξία στα κράτη-μέλη για να προσαρμοστούν στις τοπικές συνθήκες. Η έκθεση του Κοινοβουλίου λέει ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να αναπτυχθεί με στόχο την βελτίωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε όμως ότι δεν ε, θα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ε, προνομιακές ε, εργασιακές διατάξεις δεδομένου ότι η οδηγία έχει οδηγήσει σε διαφορές μισθών και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν θα πρέπει επίσης να οδηγηθούμε σε παράνομες πρακτικές. Θα πρέπει από κοινού να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλο τον τομέα ανεξαρτήτως του καθεστώτος, του εργασιακού τους καθεστώτος. Ξέρουμε επίσης ότι ε, οι αγορές online είναι σημαντικός παράγοντας πλέον. Ε, οπότε ε, η έκθεση αυτή που αναφέρεται και σε αυτό είναι πάρα πολύ καλή. Θέλω να την υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Φαντεκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ καταρχάς να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή Μάρκους Φέρμπερ αλλά και τους κοιόδης εισηγητές τη Επιτροπή Μεταφορών. Να τους ευχαριστήσω, λέω, για το έργο του, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκη, που εκπροσωπεί απόψε τον αρμόδιο επίτροπο και το κάνει με τρόπο πάρα πολύ επαγγελματικό, πρέπει να πω. Είναι λίγο περίεργο ίσως σε αυτή την ψηφιακή εποχή και κόσμο που ζούμε να ε, συζητάμε για κλασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Τους ε, τελευταίους μήνες έμαθα όμως ότι οι κλασικές παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες και γενικώ οι υπηρεσίες του ταχυδρομείου για πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη είναι εξαιρετική σημασία. Και δεν μιλώ μόνο για τους ηλικιωμένους, δεν μιλώ μόνο για ανθρώπους που ζουν σε αεροκατοικημένες περιοχές, αλλά ο καθένας πραγματικά ε, παραγγέλνει ε, εμπορεύματα που έρχονται με το ταχυδρομείο. Και επίσης Έχουμε και την οδηγία για την αποστολή των ταχυδρομικών δεμάτων που και με το ηλεκτρονικό εμπόριο ξέρουμε ότι είναι μια τεράστια θούσα. Ε, οικονομία. Θα ήθελα τώρα, μια που έχω το λόγο, να σας παρακαλέσω και να σας ρωτήσω μήπως μπορείτε να ψάξετε να βρείτε πόσες εκθέσεις εφαρμοστικές έχει ε, κάνει το Κοινοβούλιο, έχει διεκπαιρεώσει το τελευταίο διάστημα. Διότι ερχόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με τεράστιες δέσμες εκθέσεων πρωτοβουλίας, είναι λέγονται αυτά στη διάλεκτο του Κοινοβουλίου. Συμφωνήσαμε όμως στην αρχή της θητείας να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή, στην υλοποίηση υλοποίηση ε, της κείμενης νομοθεσίας. Ε, υπήρξε ε, μια μεγάλη ιστορία αυτή του Γέρζι Μπούζεκ για τις οδηγίες, μάλλον για τις εκθέσεις για την εφαρμογή κάποιων οδηγιών και θα ήθελα να το αναγνωρίσετε και εσείς δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα εκεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγιάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι κύριε Φέρμπερ για αλλαγή που θα υποστηρίζαμε απολύτως την έκθεσή σας γιατί είναι πολύ ισόρροπη και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ανατρέπει διότι μας μιλάει για ένα κανονισμό με τον οποίο διαφωνούμε. Δηλαδή, η έκθεσή σας και σας συγχαίρω για αυτή είναι εξαιρετική, αλλά τη διαβάζουμε υπό το φως του νέου κανονισμού για τα δέματα που μας εξαγγέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έρθει νωρίτερα Αφού τα ξέρατε τόσο πολύ, τι κάνατε με τις προθεσμίες, γιατί δεν τις στηρείτε, γιατί δεν κάνετε διαβούλευση και δεν καταδέχεστε να περιμένετε να ακούσετε το κοινοβούλιο. Γιατί σας έχει πιάσει τέτοια πρεμούρα, δεν καταλαβαίνω. Κάποιο λόγο θα έχετε μάλλον και όχι πολύ καλό. Δεν καταλαβαίνω γιατί εξισώνονται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και αποστολή δεμάτων με το roaming. Τι δουλειά έχει το roaming και οι τηλεπικοινωνίες με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τα δέματα. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα ήθελα επίσης να ζητήσω ρητά σε κάποια από τα θέματα να ξέρετε ότι θα συγκρουστούμε, θα μα βρείτε απέναντι στη μάχη αυτή με την πρόταση που φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φέρμπερ έκανε μια καλή έκθεση, ισόρροπη, τον ευχαριστούμε ε, και μάλιστα δέχθηκε και όλε μα τι τροπολογίε που προσπαθούσαμε και πάλι κάπω να διατηρήσουμε κάποια στοιχειώδη συνοχή και ε, την υπεράσπιση τη καθολική ταχυδρομική υπηρεσία με αξιοπρεπείς θέσεις εργασία. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Thank you, President, colleagues. I'd like to thank... Uh, Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και ο Σφέρμπερ για την αφοσίωσή του σε αυτή την μακροχρόνια οδηγία. Φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουμε όμως καταλήξει σε κάποια κοινή συνεννόηση. Το βασιλικό ταχυδρομείο ανάγεται σε εμά από τον, στον Ρίκο τον 8ο, τον αρχικό Brexiter. Από τότε έχει ξεκινήσει και έχει ανοίξει ο τον αρχικο brexiter απο τοτε εχει ξεκινησει και εχει ανοιξει ο για ενοποιημένη ταχυδρομική υπηρεσία στον Ρωμαίο Βασίλειο με τους ταχυδρόμους κλπ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά που έχουμε εμείς από το 2011 πηγαίνουν πολύ πέρα αυτά που λέμε εδώ για καθολική υπηρεσία. Υπηρεσίες ε, για τα άτομα, δέματα κτλ. Δυστυχώς, λόγω λοιπόν της κοινωνικής διάστασης και τη περίληψή τη δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τον εισηγητή. Όχι επειδή δεν υποστηρίζουμε τις ευκαιρίε και τις, συνθήκες, τις καλές συνθήκες αλλά στην παράγραφο 48 για τους ε, ταχυγράφους στα οχήματα το 14 μετά από εκτονή συζήτηση για την περίληψη αυτών των οχημάτων καταφέραμε τελικά να δώσουμε στήριξη. Και τώρα, Πρόεδρε, ζούμε σε ένα κόσμο που όλοι μας αγοράζουμε online αγαθά και αναμένουμε μια υπηρεσία σε 24 ώρη βάση. Έχουμε νέες μορφές επιχειρηματικότητας σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό κύριε ε, Φόρπε δεν υποστηρίζω την έκθεσή σας εκτός και αν αποσυρθεί 48 και ελπίζω αυτό να συμβεί μέχρι αύριο στην ψηφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελίτσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε αφορούν την επικοινωνία και δεν νομίζω να έχει αλλάξει και τίποτα ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα της επικοινωνίας. Ποια είναι αναλογία μεταξύ Facebook, WhatsApp και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Είχε αλλάξει θεματικά αυτή η αναλογία. Και νομίζω ότι αν κοιτάξουμε το παρελθόν σε αυτό καταδεικνύει. Πάντως ο συνάδελφος Φέρμπερ δεν ακούσε στενά την οδηγία, είχε ένα πιο ευρύ και ανοιχτό πνεύμα να, να εξετάσει δηλαδή, τις μελλοντικές εξελίξεις. Νομίζω προς τα εκεί πρέπει να βαδίσουμε, να δούμε τους κατανοητές και να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις τους. Για μένα καλύτερος τρόπος θα ήταν να έχουμε ένα σταθερό κανονιστικό περιβάλλον με υψηλή ποιότητα, καθολικές υπηρεσίες και με κάποιο βαθμό ευελιξίας με ανεξάρτητες, το τονίζω ανεξάρτητες εθνικές αρχές που θα επιτηρούν την κατάσταση στην αγορά αλλά να έχουμε ένα σταθερό ξαναλέω περιβάλλον μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν μακρόχρονη παρουσία στην αγορά και των νέων επιχειρήσεων, τη επιχειρήση καθολικού χαρακτήρα όπω και τι άλλε ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει και έχουμε επίση και μία συνειδητοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει η διασυνοριακή ε, συνεργασία. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, όχι ο προστατευτισμό που συναντάμε σε κάποιε χώρε. Για μένα πρόκειται κυρίε και κύριοι για μία αρχή. Αναμένουμε την επόμενη πρόταση, ο αντιπρόεδρο ήδη το ανέφερε, για την παράδοση δεμάτων και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Προσβλέπω σε αυτό και ελπίζω να ακολουθήσουμε τις αρχές για τις οποίες συμφωνήσαμε στην έκθεση. Κύριε Φέρβος, ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία που είχαμε. you, Mr. Ε, ευχαριστώ κύριε Ταρίτσκα. Κονθάλεφ Πένιας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και σε άλλους τομείς η Κομισιόν κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την φιλευθεροποίηση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα επιχειρήματα αυτής της στρατηγικής είναι η διασφάλιση προσβασιμότητας όλη την Ένωση, η διασφάλιση κριτηριών ποιότητας και η προώθηση του δυναμισμού και της ποιότητας των, της απασχόλησης. Όμως τα κριτήρια και οι στόχοι αυτοί δεν τηρήθηκαν. Κάθε άλλο, οι χώρες που πιο έντονα εφάρμοσαν τις αρχές οδηγίες βρίσκονται στην αντίθετη κατάσταση. Δηλαδή με μια υποχώρηση της ποιότητας άνοδο των παραπώνων σε σχέση με τις υπηρεσίες των νέων παρόχων. Με αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητα και καθολικότητα. Οι νέοι επιχειρηματίες, οι νέες επιχειρήσεις επικεντρώνονται στις πιο επικερδείς, επικερδείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών εις βάρος των μικρών χρηστών και οι μεγαλύτερες απώλειες ε, ποιότητας εμφανίζονται στις λιγότερο συνδεδεμένες περιοχές και στις πιο αραιοκατοικημένες. Αν δούμε και τις επιπτώσεις στα εργασιακά, βλέπουμε γενικότερη υποχώρηση της απασχόλησης, μείωση των μισθών και υποχώρηση θεαματική των εργασιακών συνθήκων. Οπότε διερωτώμεθα πότε θα φτάσει η κατάλληλη στιγμή όπου τα ευρωπαϊκά όργανα θα αποδεχτούν ότι έχουν συμβεί όλα αυτά και θα εγκατελείψουν την ιδέα ότι η φιλελευθερωποίηση αποτελεί την ε, λύση για τα πάντα. Είναι κάτι το οποίο έχει αποτύχει. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώ στι δημόσιε υπηρεσίε και στην απασχόληση ποιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εύαν είναι η επόμενη ομιλήτρια. μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρμπερ, τον εισηγητή, για την έκθεσή του και για τις ε, τροπολογίες που υποβάλαμε <clears throat> οι πράσινοι. Θα στηρίξουμε την έκθεση αυτή αύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατηθούν αυτές οι καθολικές ε, υπηρεσίες ε, σαν τις ελάχιστες υπηρεσίες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να υπάρξει περισσότερη ευελιξία στο εσωτερικό των κρατών μελών έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ειδικέ ανάγκες, έτσι ώστε να είναι Βιώσιμη η υπηρεσία. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικούς τομείς προσφοράς υπηρεσιών σε ένα τομέα που η ψηφιακή τεχνολογία παίρνει όλο και περισσότερο ε, χώρο. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση όμως να υποστούν διακρίσεις οι άνθρωποι που ζουν στην Ήπεθρο σε σχέση με αυτούς που ζουν σε αστικές περιοχές και σε μεγαλοπόλους όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές. Στην έκθεση διαβάζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν εξωπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβέ να υπάρχει χρόνος ανάπαυσης και ασφάλεια για τις μεταφορές των εργαζόμενων στον τομέα αυτό. Επίσης, στην περίπτωση των διασυνοριακών υπηρεσιών υπάρχει ομαλή υπηρεσία καθώς και λογικό κόστος, το οποίο είναι κάτι το αυτονόητο, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέλη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Φέρμπερ για την εξαιρετική του εργασία. Τεκμηριωμένη μεθοδική και ο ίδιος ήταν πρόθυμος να ε, δεχτεί και τις δικές μας τροπολογίες. Επί της ουσίας πρέπει να σας πω ότι όντως ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει εδαφός, αλλά για να πετύχουν αυτές οι υπηρεσίες χρειάζεται η παραδοσιακή υπηρεσία του ταχυδρομείου, γιατί όταν παραγγέλνεις κάτι ε, online κάποιος πρέπει να στο φέρει. Επίσης σε πιο απομακρυσμένε περιφέρειες, στι πιο αεροκατοικημένες στην Ήπεθρο, το ταχυδρομείο παίζει πρωταρχικό ρόλο. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ευελιξία μα. Χαίρομαι λοιπόν που το έγγραφο τα λαμβάνει αυτά υπόψη και ιδιαίτερα ακριβώ τι τοπικέ ε, ιδιαίτερότητε και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη καλύτερα στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τις ε, διασυνοριακές ταχυδρομικές υπηρεσίες πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρέπει να έχουμε τιμές προσιτές ε, και τιμολόγηση που να καθορίζεται με διαφάνεια. Γιατί ξέρουμε ότι παραμένουν μεγάλα τα προβλήματα ε, του κόστους των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Υπάρχουν και νέες τεχνολογίες Έχουμε ακούσει ότι για την παράδοση χρησιμοποιούνται πλέον drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ε, αν αυτό προχωρήσει θα είναι πολύ αποτελεσματικό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριος Δεμόντε, για ένα λεπτό. Η κυρία, συγγνώμη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το δικαίωμα μετάδοσης και λήψης επικοινωνιών είναι ένα δικαίωμα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν μια υπηρεσία καθολικού χαρακτήρα με ψηλή προσβασιμότητα και ποιότητα. Ο όσον αναφορά τη συλλογή και παράδοση του ταχυδρομείου Στι πιο μακρινέ και αρκοτικημένε περιοχέ χρειάζεται αυτό ιδιαίτερα τη στιγμή που η παροχή αυτή τη υπηρεσία σε αυτού του τόπου είναι βασική σημασία για λόγους κοινωνική συνοχή. Δεν θα πρέπει μόνο εκτάκτο να υπάρχει ένα περιθώριο ελαστικότητα για τη διατήρηση τη υπηρεσία αυτή. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ε, εξελίξει αγορά και στι ανάγκε των χρηστών. Όμω υπό τον όρο ότι δεν θα υποχωρήσουν η ποιότητα και ο χαρακτήρα τη καθολική υπηρεσία που έχει κυρίω δημόσιο χαρακτήρα. Εξίσου σημαντικό είναι και ο ρόλο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα πρέπει να τα δραματίσουν εδώ, προσφέροντα μια ισορροπία μεταξύ ευελιξία και δικαιώματο στην πληροφόρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βοτόψκη. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αγορά των ταχυδρομικών ε, υπηρεσιών σήμερα έχει αλλάξει σημαντικά. Υπάρχουν βασικές υπηρεσίες του παρελθόντος που σήμερα πλέον δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Και βεβαίως η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι ποιες θα είναι οι νέες υπηρεσίες που θα συνεχίσουμε να χρειαζόμαστε. Κάποιοι από τους φορείς που σήμερα δραστηριοποιούνται δεν θα μπορέσουν σίγουρα να δέξουν το επιπλέον κόστος, της επιπλέον δαπάνες, διότι βλέπουμε ότι η αγορά των ψηφιακών υπηρεσιών Σίγουρα χρειάζεται ρύθμιση που θα επιτρέψει να μειωθεί το σημερινό κόστος, έτσι ώστε να μπορέσουν και νέοι φορείς και νέες επιχειρήσεις να διεισδύσουν στην αγορά. Αυτό που πρέπει είναι να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και το κόστος και την παρεχόμενη υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει η κυρία Κίλαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες αυτές που έχουν καθολικό χαρακτήρα. Θα πρέπει βεβαίως να ορίσουμε με προσοχή για ποιες ακριβώς υπηρεσίες ε, ε, σε ποιε ακριβώ υπηρεσίε θα αναφερόμαστε, ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών που πρέπει να παρέχεται σε όλους όπου και αν διαμένουν. Και βεβαίω οι διακρίσει είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε. Είναι πολύ σημαντικό οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να είναι οικονομικές, να είναι βιώσιμες και να είναι υπηρεσίες ποιότητας. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν δαπάνη, σαν άχθος. Είναι καθοριστικές για τη λειτουργία μιας κοινωνίας. Και οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ αξιόλογοι και πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντόρφμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπογραμμίζει τη σημασία της καθολικής υπηρεσίας. Η ποιότητα ζωής όχι μόνο σε αστικές περιοχές, εκεί που ζουν οι περισσότεροι ε, άνθρωποι, θα πρέπει να δώσουμε σημασία και στην Ήπεθρο και στις πιο αεροκατοικημένες περιοχές. Είναι σημαντικό να δούμε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ε, καταστάσεις και το 20% του πληθυσμού θα μπορούσε να αποκλειστεί από αυτές τις καθολικές υπηρεσίες σε κάποιες περιοχές όπως τη δική μου και αυτό βεβαίως θα είχε σημαντικές επιπτώσεις 116 κοινότητες γιατί μόνο ελάχιστες θα μπορούν να συνεχίσουν να εποφελούνται από αυτές τις καθολικές υπηρεσίες. Για τους υπόλοιπους, τις υπόλοιπες κοινότητες θα πρέπει να υπάρχει ταχυδρομική υπηρεσία μία φορά κάθε δύο ή τρεις μέρες. Φανταστείτε να πούμε ότι κάπως έτσι θα γίνει και για το τηλέφωνο, για τον τύπο, είναι σαν να μου λέτε ότι θα αρκεστούμε σε εφημερίδες οι οποίες θα είναι χτεσινές ή προχτεσινές. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Πρόκειται για μια δημόσια υπηρεσία και θα πρέπει οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να ενισχυθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να πω και εγώ ότι όντω το ταχυδρομείο είναι μια δημόσια υπηρεσία και χωρίς πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία μια συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού αποκλείεται. Και αυτό θα θέλαμε να αποφύγουμε. Να θυμόμαστε ότι αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι η πρόσβαση, η γεωγραφική εξυπηρέτηση και η οικονομική πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάποιο κόστος υπάρχει, θα πρέπει να το αναλάβουμε. Και αυτό βεβαίως συμβαδίζει και με τις προϋποθέσεις, τις απαιτήσει για την ποιότητα. Δεν θα πρέπει να μας φοβίζει ο άγριος ανταγωνισμός. Συνέβη αυτό σε μας στην Πολωνία, μειώθηκαν οι τιμές και είχαμε παροχή υπηρεσιών αυτού του είδους μέσω φούρνων ή άλλων καταστημάτων και οι υπηρεσίες ήταν τελικά κακές επειδή προσπάθησαν να εξοικονομήσουν και να περιορίσουν τα κόστη. Πρέπει λοιπόν να δούμε καταρχά τι γίνεται με το θέμα τη εργασία και ποιότητα και εδώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που υπόθηκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι από μια περιοχή της Κονόλης Υπέθρια. από την Ήπεθρο μάλλον, συγγνώμη. Και έχουμε μισό εκατομμύριο κατοίκων που δικαιούνται το μέγιστο επίπεδο χρηματοδότηση από την Ένωση. Είναι αεροκατοικημένη και απομακρυσμένη περιοχή. Οπότε οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε είναι ζωτική σημασία. Έχουμε και την νομοθεσία του 2011 στον Ηνωμένο Βασίλειο για αυτέ τι υπηρεσίε και χαίρομαι που βλέπω εδώ είμαστε κάπου στη μέση σε σχέση με διασφάλιση αυτής τη υπηρεσία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά ας μην παραβλέψουμε αυτές τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζει αυτή η νομοθεσία. Θα πρέπει οι πάροχοι αυτής της υπηρεσίας να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις μεταβολόμενες συνθήκες μετά από την μεταβολή και τη ζήτηση. Δεν χρειάζεται να έχουμε περισσότερα βάρη που θα τους επιβάλλονται μέσω περαιτέρω νομοθεσίας. Οι ψηφόροι μου λοιπόν στην Κονουάλη απορρίπτουν αυτές τις τακτικές, περιοριστικές πρακτικές, ταχογράφη κτλ. Ευχαριστώ. Η κυρία δεν είναι στην αίθουσα. Ελπίζω να έρθει αργότερα και θα της δώσουμε το λόγο όταν επανέλθει. Η κυρία έχει το λόγο. Είναι παραπάνω από ανταγωνισμό αυτό που διακυβεύεται. Θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι οι πελάτε. Και για να έχουμε ικανοποιημένου πελάτε, χρειαζόμαστε εργαζομένου που να ε, λειτουργούν ε, υπό όρου ε, αξιοπρεπή. Και η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων συμφώνησε πάρα πολύ και υποστήριξε τις δικές μας θέσεις στη γνωμοδότησή της και κατάλαβε και η Επιτροπή Μεταφορών ότι χρειάζεται αυτή η κοινωνική διάσταση και το βάλανε στην έκθεση. Γιατί πολλέ φορέ πληρώνουν τα σπασμένα του ανταγωνισμού οι εργαζόμενοι, άνδρε και γυναίκε. Εμεί ζητούμε δίκαιε, αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία ανεξαρτήτω του είδου τη απασχόληση. Γιατί βλέπουμε και πολλού αυτοαπασχολούμενου να εργάζονται και ε, σε υπεργολαβίες και σε αλυσίδες ε, προμηθευτών που ε, είναι πολύ κακές οι συνθήκες κοινωνικές. Αυτό που θέλουμε είναι ποιοτικέ θέσει εργασία και καλές προδιαγραφές για το μέλλον. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κανονικά το λόγο έχει η κυρία Ζητνιάσκα. Για να λεπτό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χάρη στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες έχει μειωθεί η αποστολή ε, ταχυδρομικών επιστολών. Παρ' όλα αυτά παραμένει μεγάλος αριθμός, 200.000 γράμματα το χρόνο ε, και δεν σημαίνει ότι χάνει το ταχυδρομείο πελάτες επειδή υπάρχει ηλεκτρονική επικοινωνία, υπάρχει και το ηλεκτρονικό εμπόριο, οπότε αυξάνονται τα δέματα. Θα πρέπει οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να είναι καθολικές, ε, αλλά οι τιμές και το κόστος που έχουμε εμείς είναι ε, υψηλότερες στη χώρα μου από ό,τι στη Γερμανία, τη Σουηδία και τα λοιπά. Δεν μπορεί το σλοβακικό ταχυδρομείο να συνεχίζει να αυξάνει έτσι τις τιμές. Και ε, θα πρέπει ε, να καλέσουμε όλους τους ενδιαφερομένους να δημιουργήσουν τις σωστές προϋποθέσεις ε, για να λειτουργεί καλά η αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Η διαδικασία Catch the Eye. Θα έλεγα ότι δεν βλέπω τον κύριο Μαριά στην αίθουσα αλλά φαίνεται ότι κατέφθασε. Ήμουν έτοιμη να πω ότι απουσιάζει ο κύριος Μαριά, αλλά καταφθάσατε κύριε Μαριά και έχετε το λόγο αμέσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες προσφέρουν ένα κομβική σημασία έργο στις αναπτυγμένες οικονομίες υπηρεσιών. Είναι ένα τομέα αναπτυσσόμενο και καινοτόμο, ο οποίο πολύ συχνά στα κράτη-μέλη αποδεικνύει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν και παραμένουν ανταγωνιστικές σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής λιτότητας. Είναι σημαντικό ότι για τις ανάγκες των πολιτών θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα σύγκλησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακάμπτονται οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όπως επιθυμεί η Επιτροπή αντίθετα η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να αξιολογείται από τους ίδιους τους καταναλωτές μέσω της διαδικασίας ενός πανευρωπαϊκού δικτύου αξιολόγησης υπηρεσιών. ποιότητα της ταχυδρομικές υπηρεσίες σημαίνει τήρηση ενός χρονοδιαγράμματος παράδοσης και παράδοσης στην ώρα. και όλα αυτά μπορούν να γίνουν. ευχαριστώ. Eh, Θα σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Η κυρία Τούν δεν επανήλθε στην αίθουσα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ντομπρόφσκη. Έχετε το λόγο κύριε Πίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, με μεγάλη προσοχή άκουσα τις απόψεις αυτών που πήραν το λόγο. Φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει η φόρος ε, οικονομική και συνεχής ταχυδρομική υπηρεσία. Όπως είπα από την αρχή, αλλάζει με ταχύς ρυθμούς η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών και φυσικά η Επιτροπή παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις. Συμφωνεί το Κοινοβούλιο ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία στην υποχρέωση για καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες ε, βάσει της ε, οδηγίας για τις ταχυδρομικές ε, υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε καλύτερη υπηρεσία και σε κάποιες από τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις και ερωτήσεις που αφορούν το σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξής. Η Επιτροπή άκουσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το οδικό χάρτη που υιοθετήθηκε το 2013 όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες τμήμα του πακέτου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα πρέπει κανείς ε, να βγάζει συμπεράσματα σε σχέση με αυτά που έγινε με την ε, οδηγία για την περιαγωγή. Εδώ ομιλούμε για τις υπηρεσίες ε, παραλαβής και αποστολής δεμάτων. Συζητούμε ήδη αυτό το θέμα στο Συμβούλιο, με το Συμβούλιο και βεβαίως θα υποβάλουμε προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Φέρμπερ, για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους πήραν μέρος σε αυτή την Επιτροπή. Δείξατε ότι έχει νόημα να ασχοληθούμε για άλλη μια φορά με το θέμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Από το 2013 ισχύει αυτή η οδηγία, έχει μεταφερθεί στην νομοθεσία όλων των κρατών μελών η δήλωση της Επιτροπής ε, όσον αφορά την ε, υλοποίηση, την εφαρμογή αυτής της οδηγίας είναι υποχρέωση της ε, Επιτροπής. Λυπούμε που οι συντηρητικοί Βρετανοί συνάδελφοι αποσύρονται <laughs> από την Επιτροπή και πολύ θα χαιρόμουν να μπορούσαν και εκείνοι να συμμετέχουν στην ψηφοφορία αύριο. Όσον αφορά τους συναδέλφους της ε, ΓΚΟΕ, έχουμε διαφορετικές ε, απόψεις όσον αφορά τις τροπολογίες. Εμείς δεν τις υποστηρίζουμε στην πολιτική μου ομάδα. Έχουμε διαφορετικές απόψεις λοιπόν. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ψηφοφορία. Πρέπει να σας πω επίσης ότι όσοι έχουν ένα δεύτερο φορέα παροχής υπηρεσιών και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα σε κάποιες ε, αγροτικές περιοχές ε, που υπάρχει και λειτουργεί δεύτερος φορέας. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε πλαίσιο. Υπάρχουν περιοχές τις οποίες όμως δεν λειτουργεί και γι' αυτό κάνω και μία έκκληση προς την Επιτροπή. Οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών εδώ θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο παντού και σε όλες τις περιοχές οι παραδοσιακές υπηρεσίες ε, στον τομέα των ε, ταχυδρομιών μέχρι τώρα ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις διασυνοριακές υπηρεσίες και όσον αφορά και τα γράμματα αλλά και τα δέματα. Ξέρω ότι σήμερα στο εσωτερικό της ε, εκλογικής μου επικράτη, περιφέρειας. Η αποστολή ενός γράμματος δεν είναι σήμερα ε, όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια και το ίδιο βεβαίως μπορεί να πει κανείς και για τις διασυνωνικές υπηρεσίες σας. Ευχαριστώ. Τέλος της συζήτησης. Αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία.